Τέτοιου είδου επομένω υψηλά επίπεδα όσον αφορά τις, τα μεγέθη αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, λέει Και τώρα. ...για την οδική ασφάλεια έληξε. Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 11.30. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του συναδέλφου Ζέιμπερ «Ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων». Θέλω πρώτα απ' όλα να παρακαλέσω τον εισηγητή, τον κύριο Ζέιμπερ, να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εξότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχά να εκφράσω τι ευχαριστίε μου προ του συναδέλφου για την επεξεργασία αυτή τη πρώτη οδηγία για την επικοδομητική συνεργασία, η οποία ξεπέρασε τα όρια των πολιτικών ομάδων, αλλά βέβαια και τη συνεργασία με το Συμβούλιο και βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερω για την υποστήριξή τη και την ταχύτατη υποβολή προτάσεων για λύσει που υποστηρίζουν όλες ε, οι ομάδες, όλοι οι εμπλεκόμενοι. Έχουμε να κάνουμε εδώ μια μακροπρόθεσμη πολιτική, μια πολιτική η οποία στόχο έχει να εξασφαλίσει για τους πολίτες μας, για τους συμπολίτε μας, καθαρό νερό. Καθαρό νερό το οποίο όμως ταυτόχρονα και η ουσία επιβίωση, είναι η βάση επιβίωση για κάθε έμβιο οργανισμό στον πλανήτη μας και έχει τεράστια σημασία ως εκ τούτου. Θα υπενθυμίσω την οδηγία πλαίσιο η οποία αποτελεί ένα έγγραφο βάση, ένα θεμελιώδες έγγραφο με πρωτοφανή ε, στοιχεία παγκοσμίω. Καταρχάς γιατί καλύπτει όλα τα ύδατα. Δεύτερον γιατί δουλεύει πέραν των συνόρων, λειτουργεί πέραν των συνόρων. Και τρίτον προβλέπει μέχρι το 2015 την καταγραφή όλων των, μάλλον την επίτευξη όλων των θετικών, των καλών αποδεκτών επιπέδων για ουσίες στα υδατά μας. Εδώ η μεγάλη σημασία της είναι ότι προσδιορίζει συγκεκριμένες χημικές προδιαγραφές και η επίπεδα χημικών ουσιών στα ύδατα σε συγκεκριμένους όρους μέχρι το 2015. Βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με την, ε, με, την προστασία του περιβάλλοντος και με την προστασία από τις χημικές ουσίες, ε, ε, και των επιφανειακών υδάτων και έχουμε να κάνουμε με προδιαγραφές ποιότητας που προτείνονται από την οδηγία αυτή με συμπερίληψη 15 νέων ουσιών. Είχαμε οδηγία του 2003 με 30 περίπου συγκεκριμένες ουσίες οι οποίες καταγράφονταν ως επικίνδυνες για το ε, νιδάτινο ορίζοντα και τον άνθρωπο και για το 2015 προτείνεται μια σαφής διαδικασία, σαφώς προσδορισμένη διαδικασία για με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να ε, αναθεωρηθούν για επτά συγκεκριμένες ουσίες τα πρότυπα ποιότητας. Αλλάζουν ωστόσο τώρα και νέες Αλλάζουν τώρα και οι μέθοδοι μέτρησης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βεβαίως επιδιώκουμε να έχουμε καθαρό νερό για τον πολίτη της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε την παρουσία στο φυσικό περιβάλλον χημικών ουσιών που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν στην κατάρτιση ενός πακέτου που έχει τα χαρακτηριστικά, έναν κατάλογο ουσιών που τίθενται υπό παρακολούθηση και οι οποίες στη συνέχεια θα ε, ε, συμπεριληφθούν σε ένα κατάλογο με ουσίες επικίνδυνες ή ανησυχητικές ή μη επικίνδυνες Άρα έχουμε αυτό το monitoring, αυτό τον κατάλογο παρακολούθησης που ξεκινάει με 10 ουσίες και θα συμπληρώνεται κάθε χρόνο με μία επιπλέον ουσία. Δεύτερον έχουμε τις λεγόμενες φαρμακευτικές ουσίες με ένα πολύ σημαντικό βήμα για τις ε, ορμόνες και το στεροειδές αντιφλεγμονώδες δικλοφενάκι το μύστερο ιδέα, συγγνώμη, αντιφλεγμονώντας την ε, που πρέπει να τεθούν υπό παρακολούθηση και άρα μπορούμε να παρακολουθούμε από εδώ και μπρο σε ποιο βαθμό υπάρχουν φαρμακευτικές ουσίες, εμφανίζονται στα ύδατά μας φαρμακευτικές ουσίες. Μέχρι το 2021 και έως το 2027 έχουμε τις ουσίες αυτές στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής με στόχο την τήρηση των προτύπων ως το 2027 και συγκεκριμένα παρακολουθούμε εάν ε, μία ουσία για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια μπορεί να έχει επιπτώσει ή να επηρεάσει την ποιότητα των υδάτων, περίπτωση κατά την οποία μπορεί να θεωρηθεί η αδειοδότηση τη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ζέμπερ. Ο κύριο Ποτότσινγκ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Καταρχήν και πρωτίστως θα ήθελα να επηρεασει την ποιοτητα των υδατων περιπτωση κατα την οποια μπορει να θεωρηθει η αδειοδοτηση τη ευχαριστω πολυ ευχαριστω κυριε ζεπερ ο κυριο ποτοτσινγκ εχει το λογο κυρια προεδρε αξιοτιμα μελη του κοινοβουλιου καταρχην και πρωτιστως θα ηθελα να ευχαριστησω και να συγχαρώ τον εισηγητή Ρίχαρτ Ζέμπερ και την ε, εκτεταμένη δουλειά που έκανε. Ευχαριστώ επίσης την Επιτροπή που υποστήριξε τη δική μας προσέγγιση. Χάρη στην υποστήριξη της Επιτροπής καταφέραμε να διατηρήσουμε τις πιο σημαντικούς στόχους στο συμβιβαστικό κείμενο των προτάσεων μετά από διαπραγματεύσεις που θα μπορούσα να τις ε, ε, χαρακτηρίσω ως θέτουσες τουλάχιστον μια μεγάλη πρόκληση. Είναι σημαντικά όλα αυτά τουλάχιστον για τρεις λόγους. Καταρχήν παρέχει μια απαραίτητη αναθεώρηση του καταλόγου των ρηπογόνων ουσιών, των ε, ουσιών προτεραιότητας που επηρεάζουν τα ύδατα. Η αναθεώρηση αυτή απορρέει από την επιστημονική έρευνα πάνω σε ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών συμπεριλαμβάνων εκείνων ε, που εντόπισε το Κοινοβούλιο όταν υιοθετήθηκε το 2008 η οδηγία ε, για τις ε, επικίνδυνες ουσίες, για τα περιβαλλοντικά πρότυπα, με συγχωρείτε. Πολλές από τις ουσίες αυτές είναι έντονα εμένουσες, ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες, τοξικές, υψηλά τοξικές ή προκαλούν διαταραχές στο ενδοκρινικό σύστημα του οργανισμού θα πρέπει να μειώσουμε τη συγκεντρώση των ουσιών αυτών σε επίπεδα ασφάλειας και θα πρέπει να, σταδιακά να αποκλείσουμε την ε, απελευθέρωση των ουσιών αυτών στα ύδατα. Θα πρέπει επίσης να είμαστε ικανοί να διαπιστώνουμε την ύπαρξη των ρηπογόνων ουσιών με ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. Δεύτερον, η πρόταση εισαγάγει ρυθμίσεις για τη βελτίωση ε, της ενημέρωσης για τη χημική κατάσταση των υδάτων, ε, έτσι ώστε το κοινό να κατανοήσει καλύτερα τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ποιότητα των υδάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος συμπλήρωσε όλη αυτή τη δουλειά ε, για την έγκαιρη ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών και στοιχείων. Τρίτον, η πρόταση περιλαμβάνει ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης ε, για την διαπίστωση ουσιών προτεραιότητας στο μέλλον. Αυτός ο μηχανισμός ε, θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση πρόσθετων ουσιών, θα αξιολογεί τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία μέσω του περιβάλλοντος. Η πρόταση αυτή λοιπόν σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Ωστόσο, οι ελεύθερες φαρμακευτικές, οι τρεις φαρμακευτικές ουσίες που προτείνει η Επιτροπή βάσει ισχυρών επιστημονικών στοιχείων ε, μεταφέρθηκαν στον πρώτο κατάλογο επαγρύπνησης. Το συμβιβαστικό κείμενο αναγνωρίζει τους κινδύνους που θέτουν αυτές οι τρεις φαρμακευτικές ουσίες και διασαφηνίζει ότι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό για τη διευκόλυνση της ανάληψης μέτρων καταπολέμησης αυτών των κινδύνων. Αλλά φυσικά στη φάση που, που διατρέχουμε, οι ουσίες αυτές δεν θα περιληφθούν άμεσα στον κατάλογο προτεραιότητας. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή και αναλογική προσέγγιση. Τώρα για άλλες ε, φαρμακευτικές ουσίες και την παρουσία τους στο περιβάλλον θα τα παρακολουθούμε αυτά μέσω της ανάπτυξης μιας στρατηγικής προσέγγισης στο θέμα. Αγαπητά μέλη, πολλή δουλειά ε, βρίσκεται πίσω από αυτήν την πρόταση ε, τόσο η επιστημονική αξιολόγηση όσο και η αξιολόγηση επιπτώσεων και αντικτύπου. Πάρα πολλοί ειδικοί και ερευνητέ από τα κράτη-μέλη ε, η Επιτροπή, οι ομάδες των εμπλεκόμενων πλευρών, οι επιστημονικές επιτροπές ε, αξιολόγησαν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και συνεισέφεραν. Τα επιστημονικά στοιχεία για τους κινδύνους από τις ουσίες αυτές δικαιολογούν έναν βραχύτερο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με αυτό που προτάθηκε αρχικά. Ε, δεν πρέπει να υπάρχουν προσχήματα για να μην προχωρήσουμε. Για να αποφύγουμε περαιτέρω καθυστερήσεις όμως, δεχτήκαμε τη συμβιβαστική συμφωνία για να εξασφαλίσουμε μια πρώτη συμφωνία. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση των προτάσεων. Η κοινή στρατηγική υλοποίηση για την οδηγία των υδάτων, γι' αυτό υπάρχει. Έχουμε εξασφαλίσει ότι, έχει, ότι θα μπορέσει να, γίνει, να γίνουν όλες οι τεχνικές εργασίες και πρόσθετες κατευθυντήριες οδηγίες θα δοθούν για την περίοδο 2013 με 2015. Είμαι πεπισμένο ότι η οδηγία αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και μέσω αυτού θα έχει και θετικό αντίκτυπο στην ε, υγεία των ανθρώπων. Ωστόσο, διάφορες αλλαγές που εισήχθησαν κατά την πρώτη ανάγνωση και τις συζητήσεις, την πρόταση της Επιτροπής, απαιτεί ε, από την Επιτροπή καθιστά απαραίτητο για την Επιτροπή να κάνει κάποιες δηλώσεις ε, για τις ουσίες προτεραιότητας και για τους σχετικούς κινδύνους. Υπάρχουν οι προθεσμίες για τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και υπάρχει και η χρήση της non-opinion clause. Ε, φυσικά ε, θα σας ε, στείλουμε το πλήρες κείμενο για την καταγραφή στα πρακτικά. Ε, στο πλαίσιο των δηλώσεων αυτών η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι θετική η έκβαση των διαπραγματεύσεων, ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και φυσικά αποδέχεται τη συμβιβαστική πρόταση. Επομένω, κύριε Ζήμπερ, αξιότιμα μέλη, σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε κύριε Επιτροπή Πρωτόζνη και τώρα οι αγωγητέ των πολιτικών ομάδων. Πρώτα πρώτα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κρίστα Κλάς για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τη συνάδελφοι. Όλοι έχουμε μεγάλη ευαισθησία προς τα ύδατα, γιατί το πρώτο, η πρώτη ε, συγκέντρωση υπογραφών από πολίτες, ξέρετε, δεν αφορούσε ούτε το ευρώ, ούτε τα χρήματα, τα οικονομικά, αλλά τα νερά, τα ύδατα, τη, βούληση δηλαδή και την, ε, τον πόθο για καθαρά νερά σε ολόκληρη την Ευρώπη τα ύδατα τα έχουμε καλύψει σε πολλούς κανονισμούς και οδηγίες και προτάσεις και έχουμε ένα πολύ καλό νομοθετικό πλαίσιο. Ξέρουμε ότι θα πρέπει ωστόσο κάθε ρήπανση των υδάτων μας να αποφεύγεται περισσότερο παρά να προσπαθούμε να την αποκαταστήσουμε γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα έχουμε να κάνουμε με μια πρόταση, ύστερα από τρει τριμερεί ε, διαλόγου και μια καλή συμβαστική λύση. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ζέμπερ, ο οποίο εκπροσώπησε επάξια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι θέσει του, τι προτάσει για νέε ουσίε, για νέε τεχνολογίε, μεθόδου ανάλυση, ε, διαχείριση. Και ξέρετε ότι υπάρχουν νέες, νέα μελήματα, ανησυχίες ή κίνδυνοι ω προς ε, ουσίες που μπορεί να προκύψουν και να ρυπάνουν το περιβάλλον και τα ύδατα ιδιαίτερα με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αυτές λοιπόν τις ουσίες τις θέτουμε υπό παρακολούθηση και είναι πολύ σωστό το ότι και οι φαρμακευτικές ουσίες εγγράφονται τώρα σε αυτήν, υπάγονται σε αυτόν τον κατάλογο ουσιών υπό παρακολούθηση. Μπορούν έτσι και να συγκεντρώνονται τα στοιχεία και να αξιολογούνται. Αλλά κύριε Επίτροπε θα πρέπει να επικαιροποιείται αυτός ο κατάλογος διαρκώς και να συμπεριλαμβάνονται οι ουσίες είτε στον κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας είτε να απαλήφονται από τον κατάλογο εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν χρειάζεται. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλούμε για πραγματική παρακολούθηση, επιτήρηση της κατάστασης. Ε, με το σεβασμό λοιπόν αυτό φτάνουμε σε μια καλή ε, μεθοδολογία για την προστασία των υδάτων. Μας ευχαριστώ πολύ. Ε, από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο συνάδελφος Αρσένης για δύο λεπτά πολύ κύριε πρόεδρε επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι ζητήσαμε σε αυτή την οδηγία και καταφέραμε να είναι τα φάρμακα μέσα στη λίστα παρακολούθησης και έτσι οι πολίτες θα γνωρίζουν τις συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φαρμάκων και η επιτροπή θα είναι έτοιμη για να ξαναφέρει το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη αναθεώρηση. αποφασίσαμε την αλλαγή και ζητάμε την αλλαγή του τρόπου ε, αδειοδότησης των φαρμάκων προκειμένου να λαμβάνονται οι πτώσεις του στο περιβάλλον. πετύχαμε να υπάρχουν αυστηρότερα όρια για τις ουσίες που έχουν ήδη χαρτιστεί ως επιβλαβείς. όμως είναι πραγματικά ντροπή για το συμβούλιο ότι χαράμισε πραγματικά μια ευκαιρία για την ευρώπη για επενδύσεις για να βγούμε από την κρίση πρακτικά στις υποδομές διαχείρισης των υδάτων μεταθέτοντας την, ημερομηνία εφαρμογής των νέων υποχρεώσεων για τις ουσίες που έχουν αναδειχθεί ως επικίνδυνες και επιβλαβείς για το 2027. Όμως γενικότερα στην Ευρώπη το νερό είναι στο στόχαστρο. Σας έχω στείλει συνάδελφοι ε, σε όλους το email σας το γράμμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών που ζητάνε τη στήριξή σας με την υπογραφή σας στο κάλεσμα εναντίον της ιδιωτικοποίησης του νερού της θεσσαλονίκης. και επίτροπε σε ένα θέμα που σας αφορά άμεσα σε εθνικό πάρκο στο εθνικό πάρκο βορείας πίνδου σε περιοχή Νατούρα... προωθείται η εκτροπή ενός ποταμού μέσα από τα σχέδια διαχείρισης γίνεται νομιμοποίηση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας ίση πέντε αναμογεννητριών. είναι πραγματικά μια ντροπή μια καταστροφή ενό εθνικού δρυμού μέσα από τα σχέδια διαχείριση και σα παρακαλώ να το κοιτάξετε με προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Αρσένη. Και τώρα από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, η συνάδελφο Γκέρλινγκ, για ένα λεπτό. Thank you. Σας ευχαριστώ. Είναι υποτριότητα για μας το να υπάρχει νερό υψηλής ποιότητας, αλλά είμαστε ρεαλιστές, τι μπορούμε να πετύχουμε και με τι χρονισμό. Εγώ πάντοτε ήμουν κατά το, ότι αυτά τα τρεις φαρμακευτικές θα πρέπει να περιεχθούν σε αυτό το κατάλογο από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν και αυτό διότι τελικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το, το κόστος που πρέπει να πληρωθεί για να καθίσει τον από αυτά και λέμε για 35 δις ευρώ σε μια 20 ετία μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο για αυτή τη δουλειά οπότε και εγώ θα πρέπει να διαφωνήσω με τον ε, επίτροπο που λέει ότι έχω διάσει τα στοιχεία στη διάθεσή του. Γιατί αν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε όλοι θα ήμασταν πεπισμένοι και όλοι θα υπερψηφίζαμε. Αλλά δεν ισχύει αυτό γιατί δεν είναι και τα στοιχεία αυτά τράνταχτα. Επίση, ε, ενώ περνάμε κρίση, το κόστος του, του, της ούλεν σε διάφορες χώρες είναι απαράδεκτο. Επομένω, ε, υπάρχει τώρα εδώ πέρα συνέπεια μεταξύ τη οδηγία για το είδωρο και άλλων νομοθετημάτων. Οπότε με μεγάλη μου χαρά μπορώ να πω ότι για αυτά τα σημαντικά θέματα είχαμε στον τριμερή διάλογο κάποιους καλούς συμβασμούς ε, αλλά βέβαια είναι απαράδεκτα τα σχετικά με την εποπτεία και τα του, τα του χρονικού πλαισίου εφαρμογή του νομοθετήματο και αυτό το θεωρώ παρά. Γι' αυτό και επιψηφίσαμε. Εστρέλα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η επιμόλυνση του υδροφορορίζοντα θέτει εν κινδύνο την ποιότητα των ποσίμων υδάτων. Είναι και, είναι και πρόβλημα αυτό και για το περιβάλλον γενικότερα, οπότε γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς θα φτάσουμε σε κάποια ισορροπία όσον αφορά το νερό στην Ευρώπη. Και είχαμε βάλει στόχο το 2015. Είπαμε θα πρέπει να βρούμε κάποιες στρατηγικές, ώστε αυτού του είδους η ρήπανση να μην υπάρχει, να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις ε, ουσίες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες για τον υδροφόρο ορίζοντα. η σχετική συμφωνία δεν περιλαμβάνει αυτές τις τρεις φαρμακευτικές ουσίες σαν ουσίες προτεραιότητας, αλλά στο στον κατάλογο, στη λίστα της εποπτείας. Της ε, καλύτερα. Οπότε υπάρχει και ο κατάλογος της παρατήρησης, οπότε έτσι μπορούμε να ασκούμε κάποια εποπτεία. Στάση αναμονής. Επίσης, να δούμε στην, ε, ποιες ουσίες θα μπουν στην φαρμακοεπαγρύπνηση και πώς θα υπάρχει και κάποιο είδους ε, αλληλεπίδραση με τα βιοκτώνα και με άλλες νομοθέσει, όπως το ΡΙΤΣ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Στέλλα και το αρχή. Ζητήσει το λόγο και φυσικά θα τον πάρουν πρώτα ο συνάδελφος Ταμπάιντι. Ευχαριστώ. Κύριε Σταμπάζη. κύριε Ποτότσνικ, ο κύριος Ζέιμπερ ξεπώνησε πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα όσον αφορά το νερό. Είναι σημαντικό και για την Ουγγαρία. Να έχουμε επομένω κοινοτικό κανονισμό. Όλα τα ποτάμια τα οποία διασχίζουν, διαβρέχουν τη χώρα μας έρχονται από το εξωτερικό. Επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει ευρωπαϊκή εποπτεία. Το 2000 είχαμε στον ποταμό Τίσα πρόβλημα με το Κιάνιο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι για την ποιότητα του νερού. Έγιναν κάποια βήματα πρώτα από το που πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν κάποιε χώρε στο νότιο τη Ουγγαρία όπου ακόμα υπάρχουν, ακόμα μολύνουν τα, τα, τα ύδατα με αζωτούχε ουσίε. Επομένω, γι' αυτό το λόγο για μα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτονομία. Obrigado, Sra. Presidente. A água é um bem público inalienável. Είναι δημόσιο αγαθό το νερό, ε, κυρία Πρόεδρε. Και επομένω θα πρέπει να θεσπίσουμε κάποια κριτήρια να τα τηρήσουμε ούτως ώστε να προστατευτεί και το περιβάλλον και η δημοσία υγεία. Όμως, εκτός από τα κριτήρια, χρειάζεται να υπάρχουν και κάποιες ε, δημόσιες κρατικές υπηρεσίες που να ασχολούνται με έρευνα ε, στον τομέα του νερού. Να έχουμε κάποιους ειδικού και να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία αυτού του δημοσίου αγαθού στρατηγικής σημασίας σε πάρα πολλές χώρες διακυβεύεται επομένω η ποιότητα του νερού και στη δική μου χώρα την Πορτογαλία διότι συνεχώς βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθάει και επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση των εταιριών υδάτων. Δεν γίνεται έτσι καλή εποπτεία της ποιότητας του παρεχομένου υδάτος. Επομένως εδώ πέρα αγόμεθα εις μία αντίφαση. Λέμε εδώ διάφορα για να διολύσουμε αυτή την νομοθεσία, αλλά από την άλλη πάμε για την ιδιωτικοποίηση μέσα από τι σημαντικέ διαμαντεύσει με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήταν εύκολες διαπραγματεύσεις, όπως ξέρει ο κύριος Ζέμπερ πάνω από 10 ομάδες εργασίας με το Συμβούλιο, τρεις τριμερείς διάλογοι, τρεις τεχνικοί διάλογοι, οκτώ συναντήσεις με την Κορεπέρ. Νομίζω πολλή δουλειά, ε, αλλά καλή δουλειά. Ε, πολύ καλή δουλειά για να γίνουν όλα αυτά ε, δυνατά και χωρίς τη βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη λίστα επαγρύπνησης, για τις φαρμακευτικές ουσίες για το θέμα του κόστους το οποίο σχολιάστηκε. Πάντοτε όταν προτείνουμε κάτι κάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου. Το ξέρετε. Και βέβαια δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Πάντα κανείς πρέπει να κοιτά και τις δύο όψεις του νομίσματος. Ποιο είναι το, κόστ, το κόστος για να επανορθωθεί μια κατάσταση και ποιο θα είναι το κόστος αν την αφήσουμε έτσι. Όταν κάνουμε την αναθεώρηση στα 5 ή στα 10 χρόνια από τώρα, σας εγγυώμαι ότι η αξιολόγηση αντικτύπου θα δείξει ότι το κόστος για την επιδιόρθωση του θέματος είναι ακόμα πιο υψηλό. Επομένω, υπάρχουν επιχειρήματα για την, να μην υιοθετούμε τέτοιου τύπου λύσεις. Πάντοτε πρέπει να ε, συγκρίνουμε το κόστος και το όφελος και πάντοτε πρέπει να προβαίνουμε σε μια στάθμιση. Ε, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά με τρόπο που να βελτιώνει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον φυσικά, αλλά με αποτελεσματικό προ το κόστο τρόπο. Ε, για τις ενδείξεις πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας βασίζονται σε ενδείξεις πάντοτε. Ε, θυμάμαι ο κατάλογος των προτάσεων ήταν πραγματικά μακρύς. Ε, σε επιστημονικές ενδείξεις λοιπόν βασιζόμαστε και φυσικά οι επιστήμονες ε, εάν επεξεργαστούν και άλλες ενδείξεις στο μέλλον πάλι θα τις λάβουμε υπόψη μας είτε προέρχονται από τον τομέα των επιχειρηματιών είτε από τον τομέα των πανεπιστημίων είτε από τον ε, τομέα των πολιτών, των εμπλεκόμενων πλευρών. Ε, θα τα λαμβάνουμε υπόψη μας πάντοτε αυτά τα πράγματα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να εφαρμόσουμε την πρόταση, να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη όσο το δυνατόν ε, στενότερα και αυτό ακριβώς σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξή σας προς την πρόταση, ε, την υποστήριξη αυτή που προσέφερε ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Ε, και τώρα ο εισηγητής Ρίχαρτ Ζέμπερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κυρία Πρόεδρε. Όπως είπα, ήταν δυνατή αυτή η επιτυχία μόνο και μόνο χάρη στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Όπω είπε και ο κύριο Επίτροπο, θα επιμένω και εγώ στην ανάγκη τη υλοποίηση, γιατί η ποιότητα αυτή τη ε, πρόταση ε, θα κριθεί από την υλοποίησή τη, από την πραγματική εφαρμογή τη. Εάν ε, κοιτάμε το κόστο τη εφαρμογή, θα πρέπει να κοιτούμε και το όφελο που θα προσφέρει αυτό το νομοθέτημα, γιατί το κόστο τη δημόσια υγεία από την ρήπανση των υδάτων είναι πάρα πολύ μεγάλο και, πολύ, και πολλαπλάσιο μάλιστα από το κόστος της εφαρμογής ε, των διατάξεων της οδηγίας. Για δε τις φαρμακευτικές ουσίες. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και ορθό βήμα και βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε να συλλέγουμε δεδομένα δεν θα απαγορευθεί κάποια φαρμακευτική ουσία λόγω της πολιτικής των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς θα είμαστε σε θέση να οργανώνουμε συστήματα συλλογής στα κράτη-μέλη και την υπεύθυνη ε, αποκομιδή φαρμάκων που δεν χρησιμοποιούνται. Και αυτό βέβαια αφορά τα φάρμακα και ε, για τον άνθρωπο αλλά και τα κτηνιατρικά φάρμακα. Και θα ήθελα να εκφράσω την ευχή και ελπίδα προς τον Επίτροπο Ποτόσνικ η Επιτροπή ως συλλογικό όργανο να παρακολουθήσει την πρόταση του Επιτρόπου Μπαρνιέ να αποκλειστεί δηλαδή να εξαιρεθεί από την οδηγία για τις ε, ε, δημόσιες συμβάσεις, ο τομέας των υδάτων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, είναι ένα πάρα πολύ, ένας πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας αυτός των υδάτων και για τον πολίτη με ιδιαίτερη σημασία και συναισθηματική και γι' αυτό θέλουμε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς ασφαλώς διατάξεις, αλλά δεδομένου ότι αυτό δεν το έχουμε επιτύχει ακόμη, θέλουμε να συμφωνήσει το συλλογικό, ο συλλογικό όργανο η Επιτροπή να αποκλειστεί το μέσο των υδάτων από τις δημόσιες συμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζέμπερ. Κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνεται η συζήτηση, η ψηφοφορία αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι παρεμβάσεις